Πάμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ας αρχίσουμε παρακαλώ. Καθυστέρησα κάπως. Γι' αυτό και θα είμαι αρκετά γρήγορος στα προκαταρκτικά. Καταρχήν ανακοινώσει του Πρόεδρου πριν να ξεκινήσουμε τη δημόσια ακρόαση. Σε ό,τι αφορά το γλωσσικό προφίλ της Υποεπιτροπής, δεν θα έχουμε σήμερα διερμηνία σε δανεικά, φιλανδικά, σουηδικά, λετονικά, σλοβενικά, μαλτέζικα, βουλγαρικά, τσεχικά, σλοβακικά και στονικά. Μην ξεχνάτε ότι τα τακτικά μέλη έχουν προτεραιότητα στη διερμηνία για τις γλώσσες τους. Μετάδοση της ακρόασης θα γίνει απευθείας από το δίκτυο του κανάλι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Καταρχήν, ο κύριος Αλμπερτίνη, ο πρόεδρος ΑΦΕΤ, μας ενημερώνει ότι στην ΑΦΕΤ θα έρθουν οι ακόλουθοι επικεφαλεί αντιπροσωπιών. Ο Χάνς Δίτμαρ Σφάισκου, το Μάρκο Σέντερε, το Λάρς Γκούναρ Βίγκεμαρκ, ο Φιλίπ Δημήτροφ, η Αντζελίνα Άικχορστ. Τη ημερομηνία θα σα τη ανακοινώσει η Γραμματεία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και το ένα το Συνέδριο Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα, που ε, οργανώνεται από τον Behörden Spiegel σε στενή συνεργασία με τον κύριο Φον Βόγκαου, τον πρώην ε, πρόεδρο της ε, Υποεπιτροπής, θα γίνει σε 9 και 10 Οκτωβρίου 2010 στο Βερολίνο. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να χρησιμοποιήσει τα, ταξιδιωτικά, τα κονδυλιά του για το ταξίδι. Και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να αποταθείτε στη γραμματεία της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το κυρίως θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι ε, ένα πολύ επίκαιρο και επικίνδυνο θέμα, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, που είναι πραγματική απειλή για τις κοινωνίες μας. Έχουμε επιφανείς και κορυφαίους προσκεκλημένους στην ε, δημόσια μας ακρόαση και θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω ορισμένους προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, ε, ενώ όσο περιμένουμε και τους άλλους. Έχουμε τον κύριο, την κυρία Ένα Κεντικ, νομικό σύμβουλο του Κέντρου Αριστείας για την ε, Άμυνα στον Κυβερνοχώρο από το Τάλιν της Εστονίας. Έχουμε τον Δόκτωρ Ούντο Χέλμπρεχτ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας ε, Δικτύου και Πληροφοριών, της ΕΝΙΣΑ δηλαδή, είναι διευθυντής, και έχουμε τον κύριο Ανδρέα Σερβίκα, από την Γενική Διεύθυνση ΙΦΣΟ για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις με τις κυβερνοεπιθέσεις. Είχαμε και τα συμβάντα στην Εστονία, είχαμε προβλήματα στη Γεωργία κατά τη διάρκεια της ρωσογεωργικής διένεξης και Γνωρίζουμε και από πληροφορίες από τις Ηνωμένε Πολιτείες πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και μάλιστα πολλές οργανώσεις ασχολούνται με το θέμα αυτό και το ΝΑΤΟ και άλλα φόρα και οργανισμοί. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ενημερωθούμε και εμείς στην υποεπιτροπή μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Ξέρω ότι οι πυρογνώμονές μας έχουν ετοιμάσει κάποιες ομιλίες με παρουσιάσεις και διαφάνειες και θα ήθελα να δώσω το λόγο, δεν ξέρω, οι κυρίες φυσικά προηγούνται, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ένεκεν Τικ από την Εστονία. Thank Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το νομικό πλαίσιο της ασφάλειας στον κυβερνό χώρο το δικό μας κέντρο αριστείας του Τάλιν θα σας παρουσιάσει την δική του άποψη. Καταρχήν να σας δώσω λίγα στοιχεία για το ιστορικό και να σας εξηγήσω και την προσέγγισή μας για τα νομικά θέματα σε ό,τι αφορά το κέντρο αριστείας μας ε, για την κυβερνοασφάλεια που έχει ολοκληρώσει μια τριετία λειτουργίας και προσπαθεί να διαμορφώσει μια γενική γνώμη για το πώς ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κυβερνοασφάλεια υπό το πρίσμα το νομικό και κυρίως υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου και όχι μόνο ε, για αυτά τα θέματα, αλλά και για θέματα ποινικά και για θέματα τηλεπικοινωνιών. Εγώ είμαι νομικός, αλλά στο κέντρο αυτό αριστείας του Τάλιν η αποστολή μου ε, είναι να κατανοήσω και να παρακολουθήσω τον αλληλοσχετισμό μεταξύ νόμου, δικαίου και πολιτικής. Γιατί υπάρχουν κάποιες ε, συνέπειες σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία που θα πρέπει να αντιληφθούμε για να ξεπεράσουμε τις ασυνέπειες μεταξύ πολιτικής και δικαίου. Θα ήθελα καταρχάς να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση των τάσεων για την κυβερνοασφάλεια και τις κυβερνοεπιθέσεις. Βλέπετε ένα φάσμα, εμείς δυστυχώς δεν το βλέπουμε, βλέπετε ένα φάσμα λοιπόν που από τη μία πλευρά έχουμε την παραβίαση εσωτερικής πολιτικής εσωτερικών κανονισμών και διατάξεων, κάτι που συμβαίνει στις εταιρείε μας και στις οργανώσεις μας καθημερινά και το διαπιστώσαμε αυτό από την αρχή της κοινωνίας πληροφορίας, από την αρχή της ζωής της κοινωνίας πληροφορίας. Και στα, δεξιά του φάσματος έχουμε το, το, κυβερν... το ε, οπλοστάσιο τέτοιων επιθέσεων στο κυβερνοχώρο. Από νομική άποψη θα πρέπει να δούμε τι καταστάσεις αντιμετωπίζουμε που μερικές φορές χρήζουν ε, διαφορετικής ε, μεθόδου οργανωτικής, νομικής ή πολιτικής για να αποκρούσουμε μια τέτοια επίθεση. Οποιαδήποτε κυβερνοσυμβάνει, κυβερνοσύγκρουση, όπου και βρίσκεται μέσα στο φάσμα, αυτό από νομική άποψη είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πού θα το εντάξουμε στο, στο φάσμα αυτό, γιατί το νομικό πλαίσιο ή η νομική τομής που θα χρησιμοποιηθούν το νομικο πλαισιο η οι νομικοι τομης που θα εφαρμοστούν για να γίνει προσφυγή σε ένδικα μέσα και να αντιμετωπιστούν τέτοιε επιθέσει, ανάλογα με το που βρίσκονται στο φάσμα και η νομική απάντηση είναι διαφορετική. Σε ό,τι αφορά τώρα το νομικό πλαίσιο τη κυβερνοασφάλεια, όπω το αντιλαμβανόμαστε τώρα, ε, περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αυτό το νομικό πλαίσιο κάποιων ε, νομικών ε, μέσων ή ένδικων μέσων το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια του δικτύου, κάποια στοιχεία από το ποινικό δίκαιο, δίκαιο ή νομικό πλαίσιο γύρω από την εθνική ασφάλεια και φυσικά και το δίκαιο από τις ένοπλες ε, συγκρούσεις. Και τέτοια στοιχεία δικαίου χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση κυβερνών επιθέσεων. Πολύ συχνά διαρωτόμαστε αν χρειαζόμαστε σε διεθνές επίπεδα επιπλέον νομικά μέσα. Και εδώ επικρατούν δύο σχολές νομομαθών. Η μία σχολή ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στο νομικό πλαίσιο που να είναι κατάλληλο να αντιμετωπίσει κυβερνοεπιθέσεις πολιτικής φύσης, όπως αντιμετώπισε η Εστονία το 2007 ή η Γεωργία το 2008 και άλλες χώρες πιο πρόσφατα. Ενώ η άλλη σχολή σκέψη λέει ότι ε, το δίκαιό μας είναι πλούσιο, έχουμε όλες τις νομικές διατάξεις που χρειαζόμαστε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες επιθέσεις στο κυβερνό χώρο. Εμείς στο δικό μας κέντρο του Τάλιν πραγματοποίησαμε μία έρευνα για το... και μία απογραφή των νομικών μέσων που έχουμε σε διεθνές επίπεδο και που είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο αριθμός αυτών των νομικών μέσων είναι γύρω στα 50. Δηλαδή, από άποψη νομικών μέσων, έχουμε μεγάλο αριθμό τέτοιων μέσων δικαιικών ή νομικών που μπορούν να καλύψουν διάφορες πτυχές ε, πληροφορίες σε τέτοια σύγκρουση στον κυβερνοχώρο. Και έχουμε 8 με 10 διεθνείς οργανώσεις που επικεντρώνονται είτε σε κανονισμούς, σε διατάξεις ή σε χάραξη πολιτικής στον τομέα αυτό. Βλέπετε στο χάρτη ότι Η άμυνά μας εναντίον τέτοιων επιθέσεων πολλές φορές ξεκινάει από τις καθημερινές δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης. Δηλαδή ξεκινάει από μια οργανωτική ασφάλεια πληροφοριών που στηρίζεται είτε σε ιδιωτικό δίκαιο ή σε νομοθετικές διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο για το ρόλο του παρόχου υπηρεσιών ε, μέσω διαδικτύου και το συνολικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Βέβαια, η κυβερνοσύγκρουση ή η φύση τέτοιων ε, κυβερνοεπισοδίων μεταβάλλεται και από αμυγός ε, ποινικά, οικονομικά αδικήματα μετατρέπει, μετακυλείται σε αδικήματα εθνικής ασφάλειας και ε, εγκλήματος οργανωμένου. Οπότε από νομική άποψη αυτό σημαίνει ότι παρόλο που έχουμε νομοθετικές διατάξεις που μας επιτρέπουν να ε, δούμε πώς θα συνεργαστούμε με τους παρόχους υπηρεσιών ή πώς θα ανταλλάξουμε πληροφορίες. Αυτά τα μέσα που έχουμε κατά ανάγκη δεν ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις ε, κυβερνοεγκλημάτων που βάλουν περισσότερο πια κατά της εθνικής ασφάλειας. Mm, let's see. it works now. So to me... Κατά τη γνώμη μου, το θέμα δεν είναι τόσο αν χρειαζόμαστε νέες νομοθετικές διατάξεις, αλλά περισσότερο το πόσο έτοιμοι είμαστε, πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε να χρησιμοποιήσουμε το ισχύο νομικό πλαίσιο και πόσο το ισχύο νομικό πλαίσιο μπορούμε να το προσαρμόσουμε σε αυτή την αλλαγή των τάσεων στα νέα χαρακτηριστικά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που από οικονομικό γίνεται περισσότερο έγκλημα κατά της εθνικής ασφάλειας. Δεν ξέρω αυτό εγώ που ανεκοκλίνει το μικρόφωνο μου συνέχεια, λέει η μιλήτρια. Αν κοιτάξουμε τις ε, διεθνείς οργανώσεις και έτσι καταλαβαίνουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το θέμα και ποιες είναι οι οργανώσεις που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα νομικού πλαισίου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Βέβαια, το κανονιστικό πλαίσιο είναι αρκετά ευρύ και δεν αναφέρεται καν στο χάρτη η ICAN ή άλλες περιφερειακές οργανώσεις που επίσης ασχολούνται με το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Πάντως, ε, χωρίς να υπησέρχομαι σε πολλές λεπτομέρειες, για να δούμε το φάσμα αυτής, αυτό το κανονιστικό, διαπιστώνουμε ότι οι διάφορες οργανώσεις έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετική ισχύ και διαφορετικές ικανότητες ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου. Ποσοτικά βέβαια οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πιο οργανωμένες και μπορεί να καλύψει όλες τις χώρες στον κόσμο. Και η νομική ρύθμιση που μπορεί να, προκαλ... να από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο γενική και πρέπει να λάβει υπόψη τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ χωρών και περιοχών σε ό,τι αφορά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Και επειδή τέτοιες ε, επιθέσεις συμβάντα βρίσκονται εξελίξει συνεχώς τον τελευταίο καιρό, αλλάζει και η διεθνή αντίληψη, η συμφωνία για το ποιε θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιοι θα πρέπει να είναι οι τομείς προτεραιότητε. Οργανισμοί όπω το ΝΑΤΟ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίσως σε καλύτερη θέση από ποιοτική άποψη να αντιμετωπίσουν τέτοιες ε, περιστάσεις γιατί μπορούν να παρακολουθήσουν καλύτερα τις εξελίξεις στην κοινωνία της πληροφορίας να ανταλλάξουν περισσότερες πληροφορίες και να εντοπίσουν τον κίνδυνο. Βέβαια δεν εκπροσωπούνται από πολλές χώρες. Σε ό,τι αφορά τον δυνητικό κύκλο των ε, φορέων της επίθεσης, ποιες χώρες ή οργανώσεις για παράδειγμα μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν κακόβουλα τέτοια λογισμικά. Οπότε, εσκεμένα δεν θα σας αναφέρω συγκεκριμένα άρθρα της ε, συνθήκης για το έγκλημα στο κυβερνοχώρο, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχει μια συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι η πιο γνωστή συνθήκη σε ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Αυτή η συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει μια διάταξη που λέει ότι όταν διακυβεύεται η εθνική τους ασφάλεια, οι χώρες δίνονται να μην εφαρμόσουν τη συνθήκη. Πάντως υπάρχει το νομικό πλαίσιο, τίποτα δεν είναι καινούριο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Απλώς θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και όλα αυτά τα νομικά μέσα. Η περίπτωση της Εσθονίας που είχαμε την ευκαιρία να την αναλύσουμε εκ του σύνεγγης και από νομική άποψη έδειξε ότι θα πρέπει ρεαλιστικά να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτή την συνθήκη του Συμβουλίου της, Επικρα... του Συμβουλίου της Ευρώπης σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας πω τώρα λίγα λόγια για το τι υπάρχει σε διεθνές επίπεδο βλέπετε ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αφορά, ενδιαφέρει έξι από τις εφτά σημαντικότερες διεθνείς οργανώσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι διεθνείς οργανώσεις δεν ασχολούνται με θέματα κυβερνοασφάλειας ή απειλής της εθνικής ασφάλειας. Ό,τι αφορά όμως το ρυθμιστικό πλαίσιο και μια πιο περιεκτική προσέγγιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Αυτή τη στιγμή που οι χώρες αντιλαμβάνονται ότι η κυβερνοασφάλεια είναι όλο και πιο δαπανηρό ζήτημα και χρονοβόρο φυσικά, όλες σχεδόν οι διεθνείς οργανώσεις αντιμετωπίζουν το ίδιο, τον ίδιο προβληματισμό. Πώς θα βελτιωθούν και πώς θα προσαρμόσουν το ρυθμιστική τους προσέγγιση ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί από αυτή η σύσσωμη η παγκόσμια κοινότητα. Μία από τις νομικές πτυχές που πολύ συχνά αμφισβητήθηκε, ε, μάλλον τέθηκε υπό συζήτηση, είναι αν, χρειαζό, αν πρέπει να αντιληφθούμε πώς ε, θα μπορούσαμε με στρατιωτικό, για παράδειγμα, τρόπο να αντιμετωπίσουμε κυβέρνα επιθέσεις. Γιατί από αυτή την άποψη, μόνο δύο οργανώσεις ε, από άποψη νομική και πολιτική πολιτικής μπορούν να, ε, να το αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί στρατιωτικά να αποκρούσει μία ένοπλη τέτοια κυβερνοεπίθεση. Ενώ το ΝΑΤΟ πολύ συχνά προβληματίζεται. Μπορούμε να συνεννοηθούμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα αποκρούσουμε μια ένοπλη κυβερνοεπίθεση. Από νομική άποψη βέβαια δεν είναι και πολύ εύστοχη αυτή η ερώτηση. Γιατί όλα τα συμβάντα, όλα τα επεισόδια επίθεση στον κυβερνοχώρο που αντιμετωπίσαμε τελευταία στον κόσμο δεν είναι στρατιωτική φύση. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν ήταν στρατιωτική φύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν θα γίνουν στρατιωτική φύση. Αλλά αυτή τη στιγμή ο στρατιωτικό χαρακτήρα είναι περισσότερο υποθετικό. Πιο σκόπιμο θα ήταν να έχουμε μια διαδικασία παρά ένα κατόφλι, ένα όριο για το τι χαρακτηρίζεται ως ε, ένοπλη κυβερνοεπίθεση. Αυτή τη στιγμή από άποψη νομικού πλαισίου όταν έχουμε τέτοια επεισόδια στον κυβερνοχώρο φορούν περισσότερο τεχνολογία. Οπότε η αντιμετώπιση τέτοιων επεισοδίων δεν γίνονται μέσω του νόμου, του δικαίου, αλλά μέσω οικονομικών μέσων πολιτικής, ε, μυστικών υπηρεσιών κτλ. Οπότε, από νομική άποψη, το δίκαιο συμπληρώνει και στηρίζει τα άλλα καθεστώτα. Γιατί όλα τα νέα επεισόδια έφεραν στην επιφάνεια νέα νομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, πώ θα προσαρμόσουμε τι διαδικασίε ανταλλαγή πληροφοριών μα στι νέε απαιτήσει, πώ θα εξασφαλίσουμε καλύτερη συνεργασία από τους παρόχους μας τηλεπικοινωνιών και πώς θα συνεργαστούμε ή τι είδους επαφές θα έχουμε με παρόχους ε, υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και άλλων χωρών. Οπότε και οι νομομαθείς θα πρέπει να αντιληφθούν τη φύση αυτής της κατάστασης και να δουν και το αρχικό πλαίσιο των κανόνων αυτών. Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, για τον εκεί οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου έχουν καθήκον ε, συνεργασίας που κατοχυρώθηκε πριν από 10 χρόνια, που θεσπίστηκε πριν από 10 χρόνια, όταν ε, στόχος μας ήταν, στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν να έχουμε μια κοινωνία της πληροφορίας που θα χαίρει της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και της αγοράς. Σήμερα όμως που αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της απειλής και της ασφάλειας, θα πρέπει να δούμε αν αυτή η απόφαση της πολιτικής ή οι νομικές διατάξεις επαρκούν για τη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα τέτοιων επεισοδίων και την απόκρουση, την αντιμετώπιση τους, σχεδόν καθημερινά έχουμε θέματα, συνηθισμένα θέματα ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά όμω το κυβερνάγκλημα και απειλές στην εθνική ασφάλεια, όσο πιο ψηλά βρισκόμαστε στο φάσμα, τόσο ε, λιγότεροι είναι και οι ενδιαφερόμενοι. Βέβαια, εγώ περισσότερο ασχολούμαι με το ΝΑΤΟ θα σας δώσω ένα παράδειγμα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ό,τι αφορά απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν και εντολή αλλά και τα μέσα στη διάθεσή τους και κοινέ φυσικά ανησυχίες για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων. Ενώ ταυτόχρονα αλλάζουμε βεϊτάσεις του κυβερναγκλήματος, έχουμε και την κληρονομιά της κοινωνίας πληροφορίας, οπότε θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας, βολής των καταναλωτών και φυσικά ικανοποίησης των απαιτήσεων της εθνικής ασφάλειας. Το θέμα της συνεργασίας με τους παρόχους του ίντερνετ ήταν χαρακτηριστικό μας ενδιαφέρει φυσικά να εξυπηρετήσουμε και τους παρόχους και να εξασφαλίσουμε νέε ε, δυνατότητε στου ε, παρόχους, αλλά με την δημιουργία των νέων ευκαιριών και των νέων δυνατοτήτων αυξάνεται και η πιθανότητα των απειλών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε πρώτα τρεις ε, ομιλητές και μετά θα υπάρχει χρόνος για ερωταπαντήσεις και μια σύντομη συζήτηση. Ε, ο Δόκτωρ ε, Χαλμπρέχτ είναι διευθυντής της ΕΝΙΣΑ και φαντάζομαι θα θελήσει να δώσει μια απάντηση σε αυτή την απειλή. Δόκτωρ Χαλμπρέχτ, έχετε το λόγο. Για να δούμε κατά πόσον εγώ αποτελώ την ευρωπαϊκή απάντηση. Θα ήθελα να σας ε, δώσω μια γενική εικόνα, εμπειρίες ε, που έχω συγκεντρώσει από τι μπορεί να κάνει η Ενίζα για αυτό το θέμα. Δεν θα θελήσω βέβαια να μπω σε τόσες πολλές ε, λεπτομέρειες όπως η προλαλήσασα. Απλά αν δούμε σήμερα τα θέματα που μας απασχολούν ε, και το τι γίνεται στο παρελθόν σε παγκόσμια κλίμακα. Υπήρχε στο παρελθόν περισσότερο το κυβερνοέγκλημα και μερικές φορές ε, αναγκαζόμαστε να πούμε ότι δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν αλλάζει η συμπεριφορά τους. Ξεκολουθεί ο στόχος να είναι πολλοί να αποκτήσουν χρήματα άλλων, ληστείες ε, και παρεμφερεί. Αν δούμε την κυβερνο κατασκοπία και αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, μόνο που τα μέσα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Σε παγκόσμια λοιπόν κλίμακα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε διάφορες χώρες ε, στον κόσμο με διαφορετικούς πολιτισμούς. Σε ορισμένες χώρες η κατασκοπία είναι αποδεκτή συμπεριφορά. Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο ε, να ε, το κατανοήσει κανείς αυτό. Αν δούμε λιγάκι τον κυβερνοπόλεμο, αν δούμε ε, πριν από πέντε χρόνια τις δημόσιες δηλώσεις, πολλές χώρες δήλωσαν ότι επιθυμούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες τους να αντιμετωπίσουν κύβερνο επιθέσεις. Έτσι λοιπόν κατασκοπία και πόλεμος, ε, κυβερνοπόλεμος και κυβερνοκατασκοπία, αυτά ξέραμε κατά το παρελθόν. Και αν δούμε τις εφημερίδες σήμερα θα δούμε ότι πράγματι μιλάμε για ένα πρόβλημα και όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια κατ' μιλάμε για την προστασία ε, των συστημάτων ε, παροχής πληροφοριών σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το θέμα της κυβερνοασφάλειας είναι το αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύου και Πληροφοριών, του ΕΝΙΖΑ. υπήρξαν κάποια συμβάντα, υπήρξε μια ε, κυβερνοεπίθεση στην Εστονία το 2007. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε σήμερα και αυτό είναι λίγο πιο επικίνδυνο, δεξιά βλέπετε ε, μια ιστοσελίδα. Σήμερα μπορεί κανείς ε, online, σε αγορές online, αλλά και σε εφημερίδες, ο πολίτης δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει κατά πόσο έχει να κάνει με μία μολυσμένη ιστοσελίδα. Έτσι λοιπόν ε, αυτή η μόλυνση με ιούς, αυτό είναι ένα είδος δουρίου ύπου όπου μπορεί κανείς ε, να χειριστεί θέματα με τηλεχειρισμό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν σημαίνει ότι κάποιος έχει ένα σερβερ ε, ο οποίος μπορεί να ε, ελέγξει ε, τους υπολογιστές που έχουν μολυνθεί. Και έτσι λοιπόν στην Ευρώπη δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο σερβερ που δίνει την εντολή προσβολής ενός υπολογιστή με ιό. Το θέμα είναι κατά πόσον, εφόσον υπάρχει νόμος, μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Εάν λοιπόν ε, σε ένα κράτος μέλος δεχθεί κανείς μια επίθεση, χρειάζεται πολλή δουλειά για να αντιμετωπιστεί η επίθεση και το θέμα είναι σε ποιες περιπτώσεις μπορούν οι πάροχοι να κόψουν το διαδίκτυο για να μην ε, διαδοθεί περαιτέρω η προσβολή με ιούς ή επιθέσεις. Υπάρχει λοιπόν μια μετατόπιση της τεχνολογίας και το μήνυμα είναι ότι σίγουρα ε, τα πράγματα δεν βελτιώνονται, δεν αλλάζει ο κόσμος. Υπάρχουν και κάποια στατιστικά δεδομένα, ε, οι διαφάνειες αυτές έχουν δημοσιευθεί και θα τα περάσω πολύ γρήγορα. Βλέπουμε διάφορα στοιχεία για τη ζημιά που έχει προκληθεί. Ε, σήμερα υπάρχουν προβλήματα κύρους, όταν δηλαδή οι επιχειρήσεις χάνουν δεδομένα, Φύγεται το κύρος τους, όταν υπάρχει κυβερνοεπίθεση σε επιχειρήσεις, στην υποδομή τους, αυτό είναι μια ζημιά. Φανταστείτε λοιπόν ε, σε ένα χρηματιστήριο ε, να προκληθεί τέτοιου της επίθεση μπορείτε να φανταστείτε τα ποσά που θα χαθούν. Σε αυτό αυτά τα στατιστικά δεδομένα βλέπετε λεπτομέρειες ε, σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις και την ε, μετατόπιση τους. Υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα επιθέσεων. Ξεκινάμε από πάνω το αποκαλούμενο phishing και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Κατά το παρελθόν μιλάγαμε για ληστείες τραπεζών. Σήμερα μιλάμε για phishing και ψάρεμα, αν θέλετε κατά λέξη μετάφραση, ποσών από λογαριασμούς πελατών. Στην περίπτωση αυτή ε, προσβάλλεται το software και ε, αυτομάτως ε, το software αυτό αναζητά άλλα software, ένα είδος δουρίου ύπου που προηγουμένως. Ε, αυτό αποτελεί πραγματικά μία απειλή. Ε, στο κάτω βλέπετε η κλοπή ταυτότητας. Εκεί μπορεί κανείς να διαδώσει στις, ε, στην Ευρώπη ε, ταυτότητες υποτίθεται για να ε, βελτιωθεί η επιχειρηματικότητα. Το θέμα όμως πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση γιατί η κλοπή ταυτότητας είναι η επόμενη επίθεση, η κυβερνοεπίθεση που μπορεί να λάβει η χώρα. Εμφανίζονται νέες τεχνολογίες. Τέταρτο από πάνω είναι σκάντα, αυτό το σύστημα ελέγχου στον τομέα της μεταποίησης. Πριν από κάποιες εβδομάδες ε, διαβάσαμε ε, στις εφημερίδες αυτή την περίπτωση του σκανδάλου του Σκάντα. Στην περίπτωση αυτή κοινοποιήθηκε τι είδους επιθέσεις μπορεί να έχει. Το θέμα όμως, ε, δεν θέλω βέβαια να σας πανικοβάλλω, το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω είναι ότι υπάρχουν πραγματικές συμπεριφορές και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε τις συμπεριφορές αυτές ε, να τις ε, προσαρμόσουμε στη σημερινή κατάσταση στον ενδεχόμενο των κυβερνοεπιθέσεων. Όταν ζει ε, κανείς ε, σε μια φυσιολογική ζωή, ε, σε ένα σπίτι, όταν φύγει κλείνει το σπίτι του, αλλά δεν έχουμε μάθει τι να κάνουμε με το διαδίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που είναι σημαντικό σήμερα είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ε, να εκπαιδεύσουμε τους νέους για το πώς θα χειρίζονται το διαδίκτυο και βεβαίως ε, ε, αν σκέπτεται κανεί φυσιολογικά μιλάμε πάλι για θέματα ασφάλειας. Εμείς ο φορέας ο Ενίζα έχει καταστρώσει αυτή την εκστρατεία της βενετία και αν δει κανεί την υποδομή που έχουμε οτιδήποτε υπάρχει αυτό το PC παραδείγματο χάρη είναι μια τεχνολογία ήδη παπαλαιωμένη 25 ετών. Ε, δεν υπάρχει η ίδια εξέλιξη στον ε, τομέα της ασφάλειας ε, όπως υπάρχει και σε άλλους τομείς στην τεχνολογία της πληροφορικής. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ταχύτητα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερη προστασία της τεχνολογικής της πληροφορικής. Όπως σας είπα προηγουμένως, η ε, πληροφορική δεν είναι θέμα εθνικό. Αν γίνει εθνικό, τότε πια είναι πολύ αργά. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν εθνικά όρια, δεν υπάρχουν σύνορα. Σε αρκετές περιπτώσεις, αν μιλάμε για την ε, ασφάλεια της πληροφορικής, αυτό ε, πρέπει να γίνει σε μεγάλη κλίμακα, σε παγκόσμιο επίπεδο. το cloud computing παραδείγματο χάρη. Εκεί υπάρχουν νέα μοντέλα ε, για τις εφαρμογές ε, της ε, πληροφορικής, πώς αυτές μπορούν να προσφερθούν στον πελάτη. Και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με θέματα ασφάλειας πληροφορικής, θέματα νομικής φύσεως. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται όλο και περισσότερο με νέα μοντέλα και η ασφάλεια πληροφορική είναι κάτι που δυστυχώ ακολουθεί εκ των υστέρων. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε φορείς στα κράτη-μέλη, έχουμε μια μεγάλη πρόκληση ε, λόγω της συνθήκης Λισαβόνας που αφορά στον ΕΝΙΖΑ ε, εμείς καλούμε να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με άλλους φορείς. Ανέφερα ε, τον ΟΣΑ και άλλους φορείς, τον ΆΙΚΑΝ. Ε, αυτό ενδιαφέρει να συνεργαζόμαστε λοιπόν με, και με τη βιομηχανία, με βιομηχανικούς κλάδους, ε, διότι η υποδομή η καθοριστική σημασία υποτομή συνήθως βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών. Άρα δηλαδή μπορεί να υπάρξει καλή συνεργασία μόνο με τη μορφή των ΣΔΙΤ και ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, ο διάλογος στον τομέα αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία. Ο οργανισμός ο ΕΝΙΖΑ μπορεί να βοηθήσει με την τεχνογνωσία του. Εμείς εξετάζουμε αυτά τα θέματα ε, δημοσιεύουμε ε, δελτία τύπου και με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, καθημερινότητά της. Και εδώ βλέπετε μια ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων μας. ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Βίκτορ να καλωσορίσω τους υπόλοιπους καλεσμένους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Αντώνη Ριάνσκι και τον κύριο Μάρκ Άρνοχαλτ. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο ε, στον κύριο Αντρέα Σερβίντα, Καλησπέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω εδώ και να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία για το τι έχει γίνει στην Ευρώπη στον τομέα της προστασίας της υποδομής κρίσιμων πληροφοριών. Θα σας μιλήσω για το τι υπάρχει, ποια είναι η πολιτική από πίσω, ε, τι κάνουμε σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το σχέδιο δράσης προστασίας των υποδομών από κρίσιμες πληροφορίες, κάτι που έχουν, με το οποίο έχουν ασχοληθεί οι συνάδελφοι που θα με διαδεχθούν και υπάρχει, έχει εκπονηθεί και το σχετικό νομικό πλαίσιο για να στηρίξει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις απειλές που θέτει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω μια γενική εικόνα για το, τις τρέχουσες εξελίξεις. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δέσμευσή της για την προαγωγή της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή ατζέντα και της ασφάλειας στην ψηφιακή ατζέντα ε, οι νέες πολιτικές συνδέονται στενά με τη δική μας δουλειά και έτσι βρισκόμαστε σε μέσα σε ένα συνεχές με τις μέχρι τώρα ενέργειες. Κάποια αριθμοί καταρχήν. Ε, πρέπει κάτι να πω εδώ. Ένα από τα ζητήματα που έχει ανακύψει από το 2006 είναι ότι όταν κινούμεθα προς τα επάνω στις ποινικέ περιοχές είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αριθμούς αξιόπιστους. Από την άλλη πλευρά τα στοιχεία που παρέχονται από τις κυβερνήσεις ή από διεθνείς πηγές, οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Αυτές οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά θεωρούνται τουλάχιστον κοινή αποδοχής από την διεθνή κοινότητα. Και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι εκπέμπουν ένα μήνυμα. Τα στοιχεία αυτά που αναφέρουμε στην ε, μελέτη αντικτύπου που ετοιμάσαμε για το 2008 ε, εκφράζουν μία ανάλυση η οποία στηρίζει την υιοθέτηση του σχεδίου δράσης ε, για την προστασία της υποδομής κρίσιμων πληροφοριών. Εδώ βλέπετε κάποιες εκτιμήσεις 10 με 20% πιθανότητα να καταρρεύσουν τα συστήματα κρίσιμων πληροφοριών. Μιλάμε για 250 εκατομμύρια δολάρια ποσό που διακυβεύεται πιο δεν έχει σημασία, ο αντίκτυπος ο οικονομικός είναι πάντοτε μεγάλος. Από οικονομική άποψη πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι δυνατόν κάτι να πάει στραβά και αυτό δεν το λέει μόνο το Οικονομικό Φόρουμ. Ε, ε, υπάρχουν τέτοιες εκτιμήσεις για το παγκόσμιο αντίκτυπο κάποιας βασικής βλάβης, ε, μίζωνος βλάβης κάποιου συστήματος κρίσιμων πληροφοριών. Είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμήθηκε ότι ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ζημίες ύψους 200 δισεκατομμυρίων αν διακοπεί για ένα μήνα η διαδικτυακή ζωή. Ε, μιλάμε πάντοτε για μείζονε ε, βλάβες. Αυτό για κάθε χώρη θα μπορούσε ε, να προκαλέσει ζημίες που ισούνται με το 1,5 1 με 1,5 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτό θα ήταν ίσως ένα κατώτατο κατόφλι, κάτω από το οποίο δεν προκαλείται κάποια σημαντική διατάραξη ή βλάβη. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κανείς εργαλεία διαδικτυακά για να διαπράξει επιθέσεις. Νομίζω ότι μπροστά μας έχουμε πάρα πολλά εργαλεία διαθέσιμα τα φράγματα παρεμπόδισης των υποψήφιων επιτιθέμενων χαμηλώνουν όλο και περισσότερο ε, το βλέπετε στο δεύτερο τμήμα της διαφάνειας. Εδώ δείχνει πόσο κοστίζει. Και αυτά είναι στοιχεία που προέρχονται από την αγορά. Δεν είναι κρυφό αυτό. Υπάρχει μια αγορά για τέτοια εργαλεία. Μπορείς να βρεις κάτι, ένα εργαλείο 50, 60 δολαρίων ή και χιλίων ή 2.000 δολαρίων για εργαλεία παραβίασης των διαδικτυακών συστημάτων. Μιλάμε για στοιχεία που προέρχονται από ε, επιθέσεις οι οποίες πυροδοτήθηκαν από χρονικές παραμέτρους και συμπεραίνει ο αναλυτές ότι ε, υπάρχουν τα μέσα για τη διάπραξη επιθέσεων ε, και αυτό είναι το ζωφερό σενάριο ίσως που έχουμε μπροστά μας τι έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το σχέδιο δράσης που σας ανέφερα το 2009. Καταρχήν ο γενικότερος στόχος είναι να δούμε πώς θα προστατευτεί η Ευρώπη από ευνίδιες ε, επιθέσεις ε, και διαταραχές μίζωνας εμβέλειας. Όλοι εξαρτώμαστε από αυτήν την πάρα πολύ εκτεταμένη τεχνολογία και τις κοινωνικές πλατφόρμες ε, οι οποίες υπάρχουν χάρη στις στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βασιστούμε σε όλα αυτά τα διαδίκτυα, τις πλατφόρμες. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει η εκτίμηση κινδύνου να καταστεί πιο συστηματικό κομμάτι της εκπόνησης αυτών των εργαλείων, των πλατφορμών, των, συστημάτων. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με ολιστικό τρόπο. Γιατί, Γιατί είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Ε, θα πετύχουμε μόνο αν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές από το χρήστη μέχρι τα σώματα δίωξης εγκλήματος, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, τους διακομιστές, ε, όλοι, όλοι πρέπει να αναλάβουν ο καθένας την ευθύνη του για τον κοινό μας στόχο που είναι όντως κοινό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ανθεκτικό και ασφαλές το σύστημα. Και μιλάμε για ανθεκτικότητα γιατί πραγματικά η οικονομική μας ζωή ε, οι οικονομικές μας συναλλαγές, η ψυχαγωγία μας, η δουλειά μας, ακόμα και οι δημοκρατικές μας συνδιαλλαγές εξαρτώνται από αυτά τα συστήματα, από αυτή την ανθεκτικότητα, από αυτές τις τεχνολογίες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι. Για να είμαστε προετοιμασμένοι όμω όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσουμε εξοπλισμό. Και για να αποκτήσουμε εξοπλισμό πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Να μην δούμε μόνο την κατάσταση ε, εκ Αντίδραση αντίδρασης στις επιθέσεις αλλά και της πρόληψης γιατί αν συμβεί κάποια διακοπή, κάποια διαταραχή λόγω κάποιας επίθεσης ή παραβίασης τότε η λειτουργία της υποδομής μας θα πέσει κάτω από το κατώτατο επίπεδο υπηρεσιών που διέπει την κοινωνία μας και θα δημιουργήσει προβλήματα για πολλά χρόνια και αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά πραγματικά σε παγκόσμιο περιβάλλον και γι' αυτό πραγματικά χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Ποιοι είναι λοιπόν οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του σχεδίου δράσης. Πρώτον, να απομακρυνθούμε να να μετακινηθούμε από σημαντικές αλλά όχι γόνιμες συζητήσεις σε επίπεδο χάραξης πολιτικής κάτω στο πρακτικό επίπεδο. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει καταρχήν να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε ορθές πρακτικές. Γιατί, Γιατί μεταξύ των 27 κρατών μελών δεν έχουμε τον ίδιο βαθμό κατανόησης, δυναμικότητας, κατανόησης, αλλά και μέσων τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον τομέα αυτό. Όπως υπόθηκε από τον δόκτορα Χέλμπρεχτ, ο δημόσιος τομέας έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει. Γιατί? Γιατί κατέχουν την τεχνολογία, την υποδομή, τη διαχείριση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία, τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και τους χαράκτες πολιτικής, την κυβέρνηση. Αυτές οι πλευρές πρέπει πραγματικά να αναλάβουν την ευθύνη τους στον πολιτικό και στο δημόσιο χώρο. Και βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να οθήσουμε τη συνεργασία μας, να συνεργαζόμαστε καλύτερα, πιο εκτεταμένα, να... Τα, τα κράτη-μέλη πρέπει καταρχήν να εξοπλιστούν, αλλά και να ασκηθούν, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην ευρωπαϊκή διάσταση, για να μπορέσουμε και εμείς να καταστήσουμε την Ευρώπη ως περιοχή πιο προετοιμασμένη αλλά να είναι και πιο έντονη η παρουσία της στη διεθνή συνεργασία, να είναι παρούσα στη συζήτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να συμμετέχει στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των διαδικτυακών συστημάτων. Ο πρώτος λοιπόν πυλώνας είναι η προετοιμασία και προετοιμασία σημαίνει πώς θα εξοπλιστεί το κάθε κράτος μέλος με ορθές πρακτικές για να αντιμετωπίσει πιθανές ε, παραβιάσεις των συστημάτων. Ε, και όπως έχει υποθεί, συστήνουμε στα κράτη-μέλη να καταρτήσουν τη δική τους εθνική δυναμικότητα, ικανότητα προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ε, τα κυβερνητικά διαδικτυακά συστήματα να προετοιμαστούν. Εύκολα λέγεται αυτό, αλλά να μην λησμονούμε ότι ήδη έχουμε και εκ μέρους του ΕΝΙΣΑ μπορούν να με διορθώσουν να κάνω λάθος, γιατί αυτοί δραστηριοποιούνται έντονα. Εξακολουθούμε να έχουμε 11 κράτη-μέλη, τα οποία απλά προγραμματίζουν κυβερνητικά αυτοποιημένα συστήματα και συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό ε, εν τέλει όταν πρέπει μια χώρα να συμμετέχει στην συνεργασία δεν υπάρχει συντονισμός σε επιχειρησιακό επίπεδο και άρα υπάρχει ένα έλλειμμα εργαλείων και δυναμικότητας για την εξασφάλιση αυτής της πανευρωπαϊκής συνεργασίας και για το λόγο αυτό πιέζουμε τα κράτη-μέλη να συστήσουν τέτοια κεντρική, κεντρικές κυβερνητικές αρχές, γιατί δεν είναι καλό μόνο για αυτούς, είναι καλό και για τη συνεργασία μας. Αν κάτι συμβεί, ε, υπάρχουν επιπτώσεις σε όλους. Το είδαμε αυτό στις επιθέσεις που έγιναν στα δίκτυα της Γεωργίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας. Η ηλεκτρονική συνεργασία είναι πολύ σημαντική γιατί μόνο μέσω αυτής αφαιρούνται και έρονται τα εμπόδια. Ωστόσο, πέρα από το δημόσιο χώρο πρέπει να υπάρχει συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο οι εθνικέ κυβερνήσεις πρέπει επίσης να έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης των κρίσεων. Ένα από τα μαθήματα που μάθαμε στην Εσθονία ε, είδαμε ότι οι πολίτες σήκωσαν το βλέμμα στην ε, κυβέρνηση, όχι στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή στον διακομιστή. Στην κυβέρνηση είναι που κοιτάζει ο πολίτη όταν κάτι πάει στραβά. Ε, πρέπει λοιπόν να οργανωθεί κάτι στο εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης και στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτευχθεί σωστή ισορροπία μεταξύ ανταγωνισμού και εθνικής ασφάλειας, όπως είπε η πρώτη ομελήτρια. Και ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το εσωτερικό των χωρών, είναι κάτι παγκόσμιο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερο μερίδιο σε αυτή τη συνεργασία. Από την άποψη τώρα της ε, ανείχνευσης, της εξυχνίασης, πρέπει φυσικά να έχουμε ικανότητες σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το υφιστάμενο χάσμα. Αυτό πρέπει να ενταχθεί το πρέπει να ενταχθεί σε μια προ, προοπτική που θα απευθυνθεί και στον πολίτη και στη μικρομεσαία επιχείρηση. Αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει και υποδομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα σας μιλήσουν οι συνάδελφοι γι' αυτό, αλλά πρέπει να φτάσουμε και σε αυτούς που είναι πιο εκτεθειμένοι. Και οι πιο εκτεθειμένοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολίτες. Αφού λοιπόν εφοδιαστούμε με εργαλεία, και εργαλεία εξυχνίασης των εγκλημάτων αυτών, πρέπει επίσης να υπάρχουν στρατηγικές για τον περιορισμό των δυσάρεστων συνοπιών. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν, να συνταχθούν πλάνα έκτακτης αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Ε, αναρωτιέται κανείς γιατί οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους απέναντι στους πολίτες τους, αλλά αυτό φυσικά δεν μπορούν να το κάνουν μέσα σε ένα κενό, απομονωμένες. Όχι. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει διάσταση της πανευρωπαϊκής συνεργασίας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω ελέγχων και δοκιμαστικών εφαρμογών αυτών των πλάνων. Υπάρχουν κάποιες πανευρωπαϊκές ασκήσεις που μπορούν να γίνουν. Ε, με χαρά μου μπορώ να πω ότι η πρώτη μεγάλης κλίμακας πανευρωπαϊκή άσκηση για την ασφάλεια θα λάβει χώρα στις 4 Νοεμβρίου και χαίρομαι πάρα πολύ που τα κράτη-μέλη ανέλαβαν την ευθύνη να το κάνουν και ζήτησαν από την ΕΝΙΣΑ να τους βοηθήσει. Ενορχίστρωσαν δηλαδή αυτό το γεγονός το οποίο θα γίνει όπως είπα στις 4 Νοεμβρίου. Αλλά για να τα κάνουμε όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιχειρησιακών εργαλείων που έχουν που έχει η κάθε κυβέρνηση. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, όλοι ασχολούν, ε, ε, έχουμε μπροστά μας αυτά τα θέματα τα οποία είναι παγκόσμια. Και αυτή η παγκόσμια διάσταση πραγματικά αντανακλάται σε αυτά που πρέπει να κάνουμε στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών ε, και να θεσπίσουμε ως ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ποιες είναι οι προκλήσεις για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ανθεκτικότητα του διαδικτύου. Αν δεν θέσουμε προτεραιότητες, θα πολλαπλασιαστούν οι πιο τοπικές, θα τις χαρακτήριζα, προσπάθειες και προσεγγίσεις. Ε, ε, θεμητό είναι ότι και τοπικά πρέπει να δρά κανεί για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα τη ασφάλεια, αλλά με την τοπική αυτή προσέγγιση υψώνονται φράγματα στο διαδίκτυο και αυτό δεν το θέλουμε. Όλα αυτά ως προς τις δραστηριότητές μας. Για μας ένα από τα εργαλεία, ε, η ενίσα δεν είναι η απάντηση ε, στις προκλήσεις, είναι μέρος της απάντησης στις προκλήσεις. Πολλά πρέπει να γίνει από το κάθε κράτος, πολλά πρέπει να γίνει και από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά βεβαίως η ενίσα μπορεί να προσφέρει βοήθεια να προσφέρει βοήθεια για να συνεργαστούν οι χώρες, να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να οριοθετηθούν οι ορθές πρακτικές και να επιτευχθεί η συνεργασία που απαιτείται για να υπάρχει αυτή η επιτυχής ε, ηλεκτρονική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι καινούρια. Να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξε... Ε, ανήγγειλε την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη και ένας από τους πυλώνες αυτής της πολιτικής είναι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια. Γιατί είναι σημαντική η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια, γιατί αν δεν υπάρχει ασφάλεια δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη έχουμε χαμηλό ποσοστό χρήσης του διαδικτύου και των ψηφιακών υποδομών και σε αυτή την περίπτωση δεν εκπληρώνονται οι προσδοκίες ε, τις οποίες γεννά η ανάπτυξη του διαδικτύου στην Ευρώπη. Αυτά ήταν με λίγα λόγια οι προτάσεις. Βλέπετε τους τρεις ε, πυλώνες, ε, η ικανότητα, η προετοιμασία ε, που βασίζεται στο τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό συναρθρώνεται με δράσεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχρόνο και τέλος καλύτερη συνεργασία και ενισχυμένο νομικό πλαίσιο για να είμαστε αποτελεσματικοί κατά την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Επίσης όμως Πρέπει να γίνει πιο ασφαλής και η πρόσβαση στο διαδίκτυο και ερχόμαστε στο περιεχόμενο εδώ. Πώς μπορούμε να, να καταπολεμήσουμε το κακόβουλο περιεχόμενο, το πορνογραφικό κτλ. Πώς θα το καταφέρουμε ε, να έχουμε πιο ασφαλές διαδίκτυο ιδίως για τα παιδιά μας. Το πρώτο, η πρώτη ανακοίνωση για την ε, ψηφιακή ατζέντα συνοδεύτηκε από μια πρόταση εξυγχρονισμού του ΕΝΙΣΑ. Για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνέβη στις 13 Οκτωβρίου και συνοδεύτηκε από μια πρόταση που θα την αναπτύξουν οι συνάδελφοι για την ε, οδηγία αντιμετώπισης των, των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών. Η πρόταση εξυγχρονισμού του ΕΝΙΣΑ είναι πολύ σημαντική γιατί ο οργανισμός αυτός θα μπορέσει να μας γνωρίσει καλύτερα, θα μπορέσει να έχει πρόσβαση σε πιο αξιόπιστα στοιχεία και αν έχουμε στοιχεία καλύτερης ποιότητας σίγουρα μπορούμε να προβούμε σε συγκριτικές αξιολογήσεις που, και συγκρίσεις που θα είναι πιο αξιόπιστες και αυτές. Αλλά ε, ε, μια καλύτερο οργανω... ένας καλύτερα οργανωμένος και εξυγχρονισμένος ενίσα μπορεί να είναι πιο ικανός για συνεργασία και να παρέχει καλύτερη στήριξη στα ευρωπαϊκά όργανα και στα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν διασυνοριακές απειλές και επιθέσεις. Με την καλύτερη συνεργα... Αν μπορεί λοιπόν εσωτερικά ο οργανισμός αυτός να, να εργαστεί καλύτερα, μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα και εξωτερικά. Μπορεί να συμμετέχει καλύτερα στη χάραξη πολιτικής να βελτιώσει τον ε, υφιστάμενο συντονισμό, ο οποίος είναι μεν υπαρκτός, αλλά είναι περιορισμένος, πρέπει να διευρυνθεί. Ιδιαίτερα από μια άποψη που θα βάλω τώρα στη συζήτηση, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι η διαχείριση κινδύνου, αλλά η διαχείριση κινδύνου μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν μπορούμε να διασπείρουμε τους κινδύνους αυτούς, να, τους, να αναθέσουμε την αντιμετώπιση τους στα μέρη εκείνα, στους φορείς εκείνους που είναι πιο αρμόδιοι, πιο ικανοί να διαχειριστούν τους κινδύνους αυτούς. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον μας ε, οριμάζει προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης ποιότητας και μιας καλύτερης ασφάλειας. Ο Άλμπρεχτ ε, το ανέφερε πολύ μεγάλος θα είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος όμως δεν πρέπει να αφαιθεί χωρίς καθοδήγηση. Νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω και βλέπετε εδώ την ιστοσελίδα μας όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Έχουμε και από άλλη Γενική Διεύθυνση εκπρόσωπο, από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο, κύριε Χάρτβικ. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για το λόγο. Μια και έχει προχωρήσει η ώρα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μην σας κουράσω άλλο. Ο τίτλο αυτή τη δημόσια ακρόαση είναι «Η καταπολέμηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο». Εμείς ε, θα σας δώσουμε μία παρουσίαση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε την παρουσίαση του κ. Χέλμπρεχτ, του Διευθυντή τη ΕΝΙΖΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Δικτύου και Πληροφοριών. Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΙΜΣΟ για την προστασία των κέριων υποδομών πληροφοριών. Και εμείς θα σας δώσουμε κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες για την διαδομή αυτή των ε, πυλώνων που σας σκιαγράφησε κάπως ο Αντρέας Σέρβιντα και να σας ε, περιγράψω μια κατάσταση που φαίνεται κάπως συγκεχημένη όταν μιλούμε για ασφάλεια του κυβερνοχώρου και την καταπολέμηση των κυβερνοεπιθέσεων. Έχουμε το θέμα της συνολικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ένα θέμα που καλύπτει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ένα τμήμα της συνολικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τι θα πει έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το θέμα αυτό. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να πούμε τις, ε, τα εγκλήματα CIA που αφορούν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ε, διαθεσιμότητα στοιχείων ε, τεχνολογίας πληροφοριών. Αυτό είναι σημαντικό θέμα όταν μιλούμε για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και έχουμε και τα παραδοσιακά εγκλήματα που χρησιμοποιούν πια τον κυβερνοχώρο και ως πρώην ε, αστυνομικός, ε, ξεματικός αστυνομίας μπορώ να σας πω ότι τα παραδοσιακά εγκλήματα περνούν πια σε ένα νέο χώρο, τον κυβερνοχώρο. Οπότε έχουμε σε αυτή την πυραμίδα τη μία πλευρά αυτά τα παραδοσιακά εγκλήματα και ε, τις επιθέσεις από την άλλη πλευρά κατά των ε, συστημάτων πληροφοριών. Το θέμα είναι ποιος είναι αρμόδιος να αντιμετωπίσει τέτοιες επιθέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, εδώ προτείνουμε νομοθετικές διατάξεις και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα απόκειται στις διεκτικές αρχές να το αναλάβουν, αλλά υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας για τις επιθέσεις. Οπότε όταν μιλούμε για ασφάλεια, αναγκαστικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις υπηρεσίες και το στρατό και όταν μιλούμε για, τις, για τον υπολογισμό μας, για, για τους υπολογιστές, για εγκλήματα στους υπολογιστές μέσω του κυβερνοχώρου και περισσότερο επιλαμβάνονται οι διοκτικές αρχές. Ο κύριος Ράντο Μυριάνσκι θα σας πει ό,τι χρειάζεστε σε ό,τι αφορά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιθέσεις των κυβερνοχώρο. Okay, good afternoon. Uh, thanks very much, Arno. Uh, I will talk about these... Εγώ θα μιλήσω για, τις, ε, για τα εγκλήματα CIA. Όταν λέμε CIA δεν εννοούμε ε, τα Αμερικανική CIA, ναι. αλλά είναι αρχικά. Είναι εγκλήματα στον κυβερνοχώρο κατά συστημάτων πληροφοριών. Πρόκειται για κάπως βαρετά δικήματα που προσβάλλουν το σύστημα κυβερνοκατασκοπία, hacking και ούτω καθεξής. Ήδη είχαμε μια συμφωνία πλαίσιο από το 2005 για τις επιθέσεις στα συστήματα πληροφοριών και τώρα υπάρχει μια νέα πρόταση. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για το ιστορικό της, για το πώς έφτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τη νέα της πρόταση. Από την υθέτηση της απόφασης πλαίσιο του 2005 είχαμε αρχικά άνευ προηγουμένου, αλλά μεγάλες, μεγάλες εμβέλειες ε, ε, επιθέσεις ε, στην Εστονία και τη Λιθουανία το 2007 και το 2008 αντίστοιχα. Θα, θα τις ακούσετε. Ιδιαίτερα η επίθεση στην Εστονία το 2007 ήταν αρκετά ζημιογόνα για την χώρα αυτή και αρκετά θεαματική. Πρόσφατα, το Μάρτιο του 2009, τα συστήματα κυβερνήσεων και κυβερνητικών οργανώσεων 103, 103 χωρών δέχτηκαν την επίθεση κακόβουλου λογισμικού κατά απόρριτων εγγράφων. Και μάλιστα και η, και η Αμερικανική πρεσβεία και πολλές Ευρωπαϊκές πρεσβείες ε, στις Βρυξέλλες υπέσαν αυτήν την επίθεση. Και όταν λέμε για κακόβουλο λογισμικό εννοούμε τους Ιού που υποχρεώνουν τον υπολογιστή σας χωρίς να μπορείτε να το ελέγξετε να κάνει πράγματα που εσείς δεν επιθυμείτε να κάνει. Τέτοιου είδου ε, κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιείται από φτουργού ε, ε, τέτοιων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Οι ιοί που προκαλούν τέτοια σημαντική επίθεση μεγάλης ευέλειας, τις αποκαλούμε τους ιούς αυτούς botnets. Και υπάρχει και το Stuxnet, θα το ακούσετε αυτό. Το Stuxnet είναι, ήταν ένας ιός που προσέβαλε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δηληστήρια πυρηνικού σταθμούς, είχαμε για το Ιράν την, την ε, αναφορά ότι πολλές εγκαταστάσεις και σταθμοί ε, προσβλήθηκαν από το Stuxnet και στους αυτούς αποκαλούμε botnets γιατί αυτοί τι είναι η τρέχουσα απειλή. Το botnet είναι ένα δίκτυο προσβεβλημένων υπολογιστών που όταν ο hacker τους χειρίζεται από μακριά μπορεί να προκαλέσουν ταυτόχρονη επίθεση σε υπολογιστές. Οπότε μπορεί κανείς να δεχτεί την επίθεση ταυτόχρονα από εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές. Οπότε το σύστημα καταραίει. Ο υπολογιστής σας ή ο σερβερ σας δεν μπορεί να ανταποκριθεί ε, ταυτόχρονα στις υποχρεώσεις του, οπότε όλες οι ε, δραστηριότητες σας σταματούν, όλες οι εργασίες που μπορείτε να κάνετε μέσω του υπολογιστή και αυτό μπορεί να κρατήσει μέρες και δεν μπορείτε να ε, πραγματοποιήσετε τις τρέχουσες σας εργασίες μέσω υπολογιστή. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αυτό το νέο, αυτή η νέα μορφή επιθέσεων μας οδήγησε σε μια ενημέρωση της απόφαση πλαίσιο του 2005. Και μάλιστα την απόφαση πλαίσιο την προσαρμόσαμε σε μια ευρύτερη συνθήκη πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης που ήταν ευρύτερη, δεν κάλυπτε μόνο τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αλλά αξιοποιήσαμε την υπάρχουσα αυτή συνθήκη. Αυτό λοιπόν ήταν το ιστορικό. Είχαμε και μια έκθεση εφαρμογής της ε, ε, απόφασης πλαίσιο για το 2005. Η έκθεση αυτή η εφαρμογής υπευλήθη το 2008 και προβλέπει αυτή η έκθεση εφαρμογής στα συμπεράσματά της ότι ενώ το διατακτικό της έκθεσης ε, προέβλεπε ότι η σημαντική πρόοδος είχε σημειωθεί στα περισσότερα κράτη-μέλη και ότι το επίπεδο εφαρμογής της απόφασης πλαίσιο ήταν καλό, Παρ' όλα αυτά, σε πολλές χώρες ε, δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η εφαρμογή. Επίσης, η έκθεση τονίζει ότι πολλές αναφιόμενες απειλές ε, επισημάνθηκαν πρόσφατα στην Ευρώπη από την ε, έκθεση, από την συμφωνία αυτή πλαίσιο, όπως ταυτόχρονες επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την, χρήση, την εγκληματική χρήση αυτών των ιών botnets. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αυτέ οι εξελίξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο καλύτερη αντιμετώπιση των νέων απειλών. Ήδη λοιπόν το 2008, επί τη βάση αυτής της έκθεση έκθεσης, ε, τη έκθεση μάλλον εφαρμογή η ε, απολογισμού τη εφαρμογή τη απόφαση πλαισίου, διαπιστώσαμε ότι τέτοιου είδου μεγάλε ευέλειε επιθέσει στον κυβερνοχώρο αποτελούν τη χειρότερη πρόσφατη απειλή, γι' αυτό και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η απόφαση πλαίσιο. Υπάρχει και μελέτη επιπτώσεων αντικτύπου που είναι προσιτή γιατί η νέα οδηγία εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε παράλληλα με την δημοσίευση της μελέτης αντικτύπου της. Η νέα πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρει ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2010. Εγκρίθηκε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τη μελέτη αντικτύπου που σας είπα, αλλά και μαζί με μια πρόταση για την ενίσχυση του ρόλου του ΕΝΙΖΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύου και Πληροφοριών. Διαβιβάστηκε το πακέτο αυτό στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα και εδώ για πρώτη φορά παρουσιάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σύνοψη αυτής της ε, απόφασης της ε, οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρώτη συζήτηση έχει προγραμματιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών το Δεκέμβριο του 2010 και μάλιστα η διαδικασία θα ξεκινήσει το 2011. Τώρα, ως προς την ουσία της πρότασης, μια και τα botnets είναι οι, οι μεγάλες δηλαδή επιθέσεις, είναι η μείζωνα απειλή σκεφτήκαμε πώς θα, θα ποινικοποιήσουμε τη χρήση τέτοιων μέσων από τα botnets για τη διάπραξη αξιόπινων ε, ενεργειών. Επίσης είχαμε το θέμα της παράνομης υποκλοπής ε, συστημάτων πληροφοριών. Ποινικοποίησαμε και αυτό το αδίκημα. Κάτι που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική απόφαση πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όμως τμήμα αυτών των παραβάσεων, αυτών των αδικημάτων που θα, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο γενικότερο τίτλο των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η νέα οδηγία έχει στόχο επίσης τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής Ποινικής Δικαιοσύνης και της αστυνομικής συνεργασίας με την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών των μόνιμων ε, ε σημείων επαφής ε, και τη δυνατότητα άμεσα αντίδρασης μέσα σε 24 ώρες. 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ώρες τη εβδομάδα. Αυτό για το άρθρο 13. Ε, αυτό το άρθρο υπήρχε και στην αρχική απόφαση πλαίσιο, αλλά η αρχική απόφαση πλαίσιο δεν απο, ε, περιελάμβανε την υποχρέωση απόκληση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Εμείς για να επιταχύνουμε την απάντηση των σημείων επαφής ε, προσθέσαμε αυτή την υποχρέωση 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα. Και μάλιστα η αντίδραση, η απόκριση πολλών χωρών στην, στο αίτημα της Εστονίας κατά την επίθεση του 2007 ήταν ένας από τους λόγους που η αντιμετώπιση των επιθέσεων ήταν ε, ελλειπής. Δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο ελπίζαμε. Γι' αυτό και θεσπίσαμε την υποχρέωση εσπευσμένης αντίδρασης. Βέβαια, δεν ήταν ρεαλιστικό να ζήσουμε το τα κράτη-μέλη να διαθετήσουν το πρόβλημα μέσα σε 8 ώρες, αλλά όταν έχουμε κατεπίγουσα περίπτωση και μεγάλης κλίμακος, θα πρέπει να μπορεί κανείς να είναι σε θέση να δει τι βοήθεια μπορεί να περιμένει από τους εταίρους του. Οπότε η υποχρέωση αυτή που προβλέπουμε είναι ε, να απαντήσουν αυτοί που έλαβαν το αίτημα, αν μπορούν να βοηθήσουν αμέσως και με ποιο τρόπο. Για να ξέρει αυτός που ζητάει τη βοήθεια, αν μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς. Μας λείπουν επίσης και γενικότερα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για το εύρος της απειλής, τέτοιου απειλής στον κυβερνοχώρο. Γιατί για το κυβερνοέγκλημα αυτό είναι πρόβλημα συνήθως. Τα γενικά στοιχεία και τα αξιόπιστα. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαδικασίες που θα προβλέπουν τη δυνατότητα συστηματικής συγκέντρωσης από τα κράτη-μέλη στοιχείων για τις κυβερνοεπιθέσεις και θεσπίζουμε την, υποχρέ... την υποχρέωση συγκέντρωση τέτοιων στατιστικών για τα κυβερνό εγκλήματα. Μόνο για τέσσερις όμως περιπτώσεις αδικημάτων. Οι τρει περιλαμβανόταν και στο, στην απόφαση πλαίσιο. Η νομική πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών, οι παρεμβολέ σε συστήματα, οι παρεμβολέ στα δεδομένα και τέταρτο πρόσφατο αδίκημα είναι η παράνομη υποκλοπή, η παρεμβολή. Τελευταίο και πολύ σημαντικό σημείο είναι η προσθήκη πιο αυστηρών κυρώσεων. Μάλιστα, ε, ζητήσαμε τουλάχιστον δύο χρόνια να είναι η ελάχιστη ποινή φυλάκιση, ενώ η, απόφαση πλαίσιο έβλεπε τουλάχιστον ένα χρόνο φυλάκιση. Και αν υπάρχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις, που είναι τρία, ε, δηλαδή όταν το αδίκημα διαπράττει στα πλαίσια ενός ε, κυκλώματος ε, οργανωμένου, όταν διαπράττεται με βάση ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για τέτοιες επιθέσεις, αν προσβάλλει μεγάλο αριθμό συστημάτων πληροφοριών ή όταν προκαλεί σημαντικές ζημίες όπως παρεμβολή ε, σε συστήματα υπηρεσιών, η προκαλεί απώλεια στοιχείων, ή υλικές ε, απώλειες. Αυτές είναι όλες ε, επιβαρυτικές συνθήκες για τη χρήση botnet τέτοιων ιών, οπότε όταν χρησιμοποιεί κανείς ένα botnet, έναν ιό δηλαδή που χρησιμοποιεί μαζικής εμβέλειας ε, κυβερνοεπιθέσεις, αυτή η περίσταση θεωρείται επιβαρυντική. Γιατί και οι ζημιές μπορεί να είναι ανυπολόγιστες και τα θύματα πολύ περισσότερα. Και η τρίτη επιβαρυντική περίσταση είναι όταν διαπράτεται ενώ ο αυτούργος κατά την ανωνυμία του. Και πολλές φορές είναι αδύνατη η έρευνα γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ο αυτούργος ή γιατί γίνεται η φαρπαγή της ταυτότητας άλλου ή διαπράττονται ε, επιθέσεις που ενοχοποιούν τρίτου που είναι τελείω αθώοι. Γιατί κάποιο που ο υπολογιστή του χρησιμοποιήθηκε για την διάπραξη μια κυβερνοεπίθεση πολλέ φορέ είναι τελείω αμέτωχο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτέ λοιπόν όλε οι περιστάσει είναι επιβαρυντικές και οδηγούν στη μέγιστη επιβολή ποινής. Αυτά. Σα εξήγησα τι είναι στην Πότνε, τι δουσιός είναι αυτό ο Πότνε που προκαλεί μαζικέ επιθέσει στον κυβερνοχώρο. Έχουμε και του ε, παραβάτε που είναι η οργάνωση που χρησιμοποιεί, αποκτά ή παράγει τέτοιο κακόβουλο λογισμικό και το διαθέτει μέσω διαφόρων μέσων. Ένα botnet κυρίως περνάει μέσω του διαδικτύου, γι' αυτό και το net μέσα, botnet. Αλλά ε, το stuxnet, ο ιός stuxnet, είναι ένας ε, ιός που χρησιμοποιείται μέσω της χρήσης USB, κλειδιών μνήμης. Οπότε στους πυρηνικούς σταθμούς ε, ε, η προσβολή έγινε μέσω προσβεβλημένων ε, κλειδιών μνήμης, USB. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Stuxnet. Αλλά εμείς μιλούμε για botnets, τέτοιους ιούς μαζικής επίθεσης. Ο bot, που είναι ο ιός του botnet μετατρέπει έναν υπολογιστή σε ζόμπι από τη στιγμή που τον ε, προσβάλλει. Τις περισσότερες περιπτώσεις εσείς δεν ε, έχετε πάρει καν χαμπάρι ότι έχει προσβληθεί ο υπολογιστή σας και ταυτόχρονα συμμετέχει σε μια μαζική επίθεση και μάλιστα ο ιός αυτός περιμένει απλώς την διαταγή του αυτούργου για να, για να, ε, για να επιτεθεί. και έχουμε και αυτούς που ελέγχουν τα botnet και που δίνουν τη διαταγή ουσιαστικά και την κήρυξη της επίθεσης. Μέσω spam, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να σταλούν αυτές οι διαταγές ε, στα mail που έχουν γίνει, στα, στους υπολογιστές που έχουν γίνει ζόμπι, υπό τον έλεγχο δηλαδή αυτών των ιών που πολλές φορές ε, στέλνουν ταυτόχρονα εκατομμύρια spam σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μπορεί και αυτά να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές, ειδικά όταν ε, στέλνονται με τόσο μεγάλα νούμερα. Αυτά τα ζόμπι υπολογιστέ λοιπόν εκτελούν αυτές τις ε, διαταγές που παίρνουν από τον ε, ελεγκτή. Όπως συνέβη στην Εσθονία. από την ίδια μέρα είχαμε μαζικές επιθέσεις από στους σερβερ υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Τρεις έχουν ε, ζητήσει το λόγο και θα ήθελα όσοι κάνουν ερωτήσεις ε, να περιοριστούν ε, κατά το μέγιστο σε δύο λεπτά. Ο κύριος Κέλαμα από την Εστονία. Το περίμενα αυτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που μας παρουσίασαν την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται στην κυρία από την Εσθονία. Μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε περισσότερο <clears throat> για τις δραστηριότητες αυτού του κέντρου αριστείας για την κυβερνοάμυνα. Ε, λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια. Ποιοι ε, συμμετέχουν, ποια κράτη, παραδείγματος χάρη και άλλα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η Κομισιόν κατέθεσε νέες προτάσεις που είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Και όπως μας είπατε, εσείς ε, προτίθεστε να έρθετε όσο πιο γρήγορα γίνεται και πάλι εδώ στην υποεπιτροπή μας. Ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Γιάνσκι, έδειξε αυτό το θέμα της, της ατομικής ευθύνης. Για μένα όμως είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι αυτούργοι, γιατί αυτό παραμένει ένα πολύ ε, δύσκολο ερώτημα. Είτε μπορούμε να αναλάβουμε ατομικά την ευθύνη. Όταν πρόκειται για τον υπολογιστή μου, αυτό είναι σαφέ. Ε, μάλλον, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Όταν κάποιο χρησιμοποιεί το όπλο μου, νομίζω εκεί είναι πιο σαφέ. Στην περίπτωση εντοπισμού του αυτούργου, αυτό ενδιαφέρει. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι αυτό που είπε ο Δ. Χέλμπρεχτ, δηλαδή η συμμετοχή των πολιτών. Συμμετοχή των πολιτών στο να υπάρχει καλύτερη αυτοάμυνα γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε και την κοινή γνώμη και δεν πρέπει αυτό τον, το πεδίο μάχης να το αφήσουμε σε ε, καταστροφικές ομάδες γιατί το διαδίκτυο κατά κύριο λόγο θα πρέπει να εκπέμπει ε, το μήνυμα της δημοκρατίας και του νόμου. Δεν πρέπει λοιπόν να θέτουμε σε κίνδυνο βασικές ελευθερίες λόγω των κυβέρνων επιθέσεων. Και τέλος το θέμα της ε, συνεργασίας. Αναφερθήκατε σε ε, προβλεπόμενα, προγραμμαζόμενα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών. Ε, αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της εξελιγμένης κυβερνοτεχνολογίας. Αυτή βέβαια είναι και μυστική, έντονα μυστική όλα τα κράτη επιθυμούν ε, να την κρατήσουν για τον εαυτό τους στο βαθμό που την έχουν. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει κάποια ε, σύγκρουση ανάμεσα στην ανταλλαγή εμπειριών, στην εξέλιξη της τεχνολογίας και παράλληλα στην εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Σήμερα εσείς πήρατε διπλάσιο χρόνο. Κύριε Νικολάεφ. Η δική μου ερώτηση έχει σχέση με τις απειλές προς το κυβερνοσύστημα. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά σε, στο hacking. Όπως ξέρετε, μάλλον το 2010 γνωρίζετε πόσες υποθέσεις ε, κυβερνοεπιθέσεων αναφέρθηκαν ε, που να σχετίζονται με hackers. Αυτό είναι ένα επίμαχο θέμα, το hacking. Και μια άλλη ερώτηση έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα που εξελίσσεται όλο και περισσότερο. Όμως αυτό που έχει σημασία από νομική σκοπιά ε, είναι όχι τόσο το να υπάρχουν κανονισμοί όσο το να εφαρμοστεί στο μέλλον η οδηγία. Εσείς ε, προτίθεστε να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την έρευνα. Γιατί πάρα πολλά κράτη-μέλη έχουν τεράστιο πρόβλημα έρευνας. Και η τρίτη μου ερώτηση έχει σύστημα με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Μήπως έτσι έχετε κατά νου ε, το να εγκαταστήσετε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να μπορεί κανείς να αποφύγει τις κυβερνοεπιθέσεις. Υπάρχει τέτοιου είδους τεχνική δυνατότητα. Η κυρία Γκόμες. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Έχοντας κατά νου τη φύση της απειλής, αυτή η νέα οδηγία πώς μπορεί να διασφαλίσει τη συνεργασία ανάμεσα στον στρατιωτικό και το ιδιωτικό τομέα για να αντιμετωπιστεί επιτυχώ η ενδεχόμενη επίθεση. Α πούμε, στο ΝΑΤΟ υπάρχει εξελιγμένη τεχνογνωσία. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία και ανάμεσα στον ιδιωτικό και το στρατιωτικό τομέα για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεση. Κύριος Έλα. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτές τις ε, νέες ε, δομές. Κοιτάξτε, όσοι ασχολούμεθαμε με το θέμα αυτό, δεν ήμασταν και παρόντε όταν συνήφθη η Συμφωνία τη Νίκη. Επρόκειτο για έναν επώδυνο συμβασμό, όπου τα κράτη δεν τον ήθελαν και πάρα πολύ, αλλά ε, ήθελαν να δεχθούν μια συμφωνία που είχε γίνει καταρχήν στην Κρήτη και μετά μια επιτροπή η οποία βέβαια μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη συμφωνία της νίκης αλλά δεν είναι απαραίτητο να το πράξει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Ε, ποια είναι η εντύπωσή σας, τα κράτη-μέλη είναι περισσότερο πρόθυμα τον φορέα ενίζα να τον ε, ενισχύσουν στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Ε, επίσης, στο σχέδιο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δούμε τον ενδεχόμενο ένταξη της ΕΝΙΖΑ ε, στα πολιτικά τεκτενόμενα, αν είχαμε μία κλίμακα ε, θα μπαίναμε στην βαθμίδα 3. Δηλαδή αυτό που μας λείπει εμάς, που δεν βλέπουμε να υπάρχει, είναι έχουμε έναν οργανισμό, τον ΕΝΙΖΑ, χρηματοδοτείται, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον συμμετέχει στις πολιτικές αποφάσεις Κομισιόν. Κατά την άποψή μου πρέπει να συμμετέχει. Και κάτι άλλο, στο μέλλον τα ερωτήματα αυτά δεν θα πρέπει να απαντηθούν μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα υπάρξει διεθνοποίηση του προβλήματος. Οι Αμερικανοί επιθυμούν ήδη τώρα να διαπραγματευτούν με εμά. Γι' αυτό λοιπόν ο οργανισμός ΕΝΙΖΑ τι ρόλο θα καταλάβει σε αυτές οι διαπραγματεύσεις και η Κομισιόν τι θα κάνει με αυτό το πρόβλημα. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν συγκεκριμένες απόψεις για, τον, ε, για τα κονδύλια του προπολογισμού, έχουν κατευθεί και προτάσεις στο Κογκρέσο. Εσείς λοιπόν πώς ακριβώς ε, σκέπτεστε τη διεθνοποίηση του προβλήματος και αν σημαίνει αυτό τι ρόλο θα διδραματίσει ο οργανισμός ε, ΝΙΖΑ. Τελευταία ερώτηση, κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ δεν είμαι μέλος της Υποπιτροπής, αλλά ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και θα μου επιτρέψει τώρα να μιλήσω ε, ρουμανικά. Γι' αυτό αν έχετε την καλοσύνη να βάλετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να αναπτύξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία στρατηγική για την ασφάλεια της πληροφορικής με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας και τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να, ε, να υποστηρίξουν την παράταση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύου και Πληροφοριών γιατί δεν αρκεί μια πενταετία. Χρειαζόμαστε πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές και χρηματοδότηση. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω και τα μέλη τη Επιτροπής ΑΦΕΤ και τα μέλη της ΕΝΤΕ να στηρίξουν την παράταση της εντολής της ΕΝΙΣΑ, του οργανισμού ΕΝΙΣΑ, ώστε τουλάχιστον να παραταθεί για μια δεκαετία. Δεύτερο σχόλιο, σε ό,τι αφορά τις κέρδες υποδομές πληροφοριών. Δυστυχώς, εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε αρκετά μέτρα για την ε, εξασφάλιση της προστασίας ε, των χρηστών. Δεν υπάρχει θέμα διαλειτουργικότητας ε, των συστημάτων κλειδιών. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπογραφών, αλλά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Αυτό και περιμένουμε με ενδιαφέρον την αναθεώρηση τη οδηγία για τι ηλεκτρονικέ υπογραφέ και τη διαχείριση της, ε, της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Θα ήθελα επίσης ε, να επισημάνω ότι σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να καθοριστεί το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η εφαρμοστέα νομοθεσία κάθε φορά. Η νομοθεσία του παρόχου υπηρεσιών, του αποδέκτων υπηρεσιών ή ισχύει δικαιοδοσία του διακομιστή των πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά την ε, Κυβερνοευρώπη 2010, για την πρώτη πανευρωπαϊκή άσκηση για την προστασία της, των κέριων υποδομών πληροφοριών που θα λάβει η χώρα τον Νοέμβριο. Μερικέ χώρε θα συμμετέχουν άμεσα, ενώ άλλε θα είναι απλώς παρατηρητές αυτή την πανευρωπαϊκή άσκηση. Πώ θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε, να ενισχύσουμε την άμυνα αυτών των χωρών εφόσον αυτέ οι χώρε παραμένουν στη θέση του παρατηρητή και δεν μπορούν να εντοπίσουν τι αδυναμίε του ε, στο σύστημα, γιατί ένα σύστημα ξέρουμε ότι μια λυσίδα έχει το σθένος της ισχύω του, του, πιο αδύναμου κρίκου της. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι οι βουλευτές δεν είναι και εμπειρογνώμονες, αλλά από ό,τι βλέπω εσείς είστε εμπειρογνώμονες, είστε ειδικοί. Λοιπόν, θα σας δώσω χρόνο να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Φυσικά δεν αναμένουμε όλοι σας να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλώ ασχοληθείτε είτε με τα ερωτήματα που σας απευθύνθηκαν άμεσα είτε με τα ερωτήματα που θα θέλατε να απαντήσετε. Η κυρία Τίκα ζήτησε πρώτη το λόγο γιατί το αεροπλάνο της φεύγει νωρίς. Θα σας ζητήσω να περιορίσετε την απάντησή σας σε πέντε λεπτά το πολύ. Κυρία Τίκ, ευχαριστώ. Καταρχήν για το κέντρο και για, για την ιστορία. Το κέντρο δεν δημιουργήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις του 2007. Ήδη από το 2003 ε, ξεκινήσαμε και πίσω από την πρόταση αυτή ε, είναι ο τρόπος που η Εσθονία ε, έχει δομηθεί ως κοινωνία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η εξάρτηση της Εσθονίας από την τεχνολογία πληροφοριών ε, καθιστά κρίσιμο το να μπορεί να προασπίζει αυτό τον τρόπο ζωής, να προστατεύεται. Επίσημα το 2008 μπήκε η Εσθονία στο κέντρο. Εγώ μπήκα το 2006 ως μέλος της επιστημονικής ομάδας που εκπώνησε την ανάλυση της ε, ε κατάστασης ασφάλειας του κυβερνοχώρου της Εσθονίας εκείνη την περίοδο. Η αποστολή του κέντρου, όπως συστάθηκε, είναι να ενισχύσει το ΝΑΤΟ και τα έθνη του ΝΑΤΟ όσο αφορά τις αμυντικές τους ικανότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κέντρο δεν παίρνει και τα πρώιμα μέτρα που χρειάζεται, αλλά δεν είναι μια επιχειρησιακή μονάδα. Είναι ένας θεσμός που ασχολείται με την ανάλυση, την ενιολογική σκέψη, τις τεχνικές ε, λύσεις, ε, ε, παρακολουθεί τα διάφορα επεισόδια που συμβαίνουν, τα μελετά και κάνει προτάσεις, διατυπώνει προτάσεις και προσεγγίσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, σήμερα έχει τρεις τρεις κυρίους τομείς με τους οποίους ασχολείται. Εγώ προέρχομαι, εγώ ε, έχω νομικό υπόβαθρο, αλλά υπάρχει επίσης η προστασία των κέριων υποδομών πληροφοριών και οι τεχνικές λύσεις, επίσης ενιολογικές συλλήψεις ε, που αφορούν τη στρατιωτική ασφάλεια. Αυτά για το κέντρο. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να θίξω σε σχέση με την ερώτηση για το οργανωμένο έγκλημα και την ικανότητα να σκέφτεται κανείς εκ των προτέρων τα μέτρα της ασφάλειας στον ε, κυβερνοχώρο. Θα έλεγα ότι η μέρος του πακέτου είναι επίσης οι νομικές και η ιδέα ότι οι νομικές και πολιτικές λύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας δεν ε, λειτουργούν, δεν αποδίδουν σε αυτό το καινούριο παράδειγμα ασφάλειας. Μιλούμε για πολλά πράγματα, για δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων, ε, για προστασία στοιχείων, ε, για συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών στον τομέα πάντοτε του εγκλήματος. Πρέπει πάντοτε κανείς να λαμβάνει υπόψη τα θέματα και τις εκφάνσεις της ε, στρατιωτικής ασφάλειας, ε, των της στρατιωτικής διάστασης. Ε, βέβαια για να κατανοήσει κανείς πώς έχει η κατάσταση στην Εσθονία πρέπει να κατανοήσει και πώς συναρθρώνεται το στρατιωτικό με το πολιτικό. Δεν σας μίλησα για μία διάσταση ε, το κέντρο σήμερα έχει οκτώ συμμετέχοντες, οκτώ έθνη που χρηματοδοτούν. Τα, την Εσθονία, την Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία. Την είπα τη Γερμανία, ναι. Και την Ισπανία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Τουρκία ε, είναι στη διαδικασία του να γίνουν μέλη. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ο Δόκτωρ Χέλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επικεντρωθώ σε ένα, θα κάνω μάλλον ένα σχόλιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και το επίπεδο εμπειρογνωσίας που έχουμε στην Ευρώπη, στην, στον τομέα, στον κλάδο της ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφοριών Νομίζω αν δείτε το 2009 θα, θα έχετε μια καλή ιδέα για τον πώς έχει ο κλάδος στην Ευρώπη αλλά και στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπήρξε μια ερώτηση για τα στοιχεία ε, Αν δείτε, αν κοιτάξετε τι συμβαίνει στην Ευρώπη θα δείτε ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα συγκρίσιμα στοιχεία. Τα περισσότερα είναι στοιχεία που προέρχονται από τις υπηρεσίες πάταξης δίωξης του εγκλήματος, τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και λίγα από την Eurostat και τις στατιστικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά συνήθως δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων εγκλημάτων ή επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Για τα συστήματα έγκυρης προειδοποίησης. Εμείς ε, από την, στον ΕΝΙΣΑ τι κάνουμε. Από τη μία πλευρά στηρίζουμε τα κράτη-μέλη, τα βοηθούμε να οικοδομήσουν, ε, ε, να συστήσουν κάποια ομάδα ανταπόκρισης σε έκτακτες περιπτώσεις που αφορούν τους υπολογιστές σε κυβερνητικό επίπεδο. Ε, ξεκινήσαμε όταν ήμασταν μόνο 15, τώρα είμαστε 27 κράτη-μέλη. Η πρόκληση είναι ότι δεν έχουμε όλοι το ίδιο επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των κυβερνήσεων. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος χρόνος. Και το πρόβλημα είναι ότι πάντοτε ο πιο αδύναμος κρίκος ε, ότι τα πρέπει να ασχολούμαστε με το πιο αδύναμο κρίκο. Αλλά όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα όταν, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δράση τη ΕΝΗΣΑ για το επόμενο έτο, θα θα προσπαθήσουμε η συλλογή στοιχείων να είναι ταχύτερη. Θα προσπαθήσουμε επίσης το πλαίσιο τηλεπικοινωνίας για την ανακοίνωση στοιχείων να λειτουργεί πιο γρήγορα, για το διαμήρασμα στοιχείων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να έχουμε ένα ρόλο στην υλοποίηση της σχετικής οδηγίας και στο μέλλον να έχουμε καλύτερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Συνοψίζοντας, έχουμε ακόμα πολύ μακρύ δρόμο να διανύσουμε. Πάντως έχουμε σε θεσμικό επίπεδο ε, τα, τις ίδιες ανάγκες ε, άμυνας και τις ίδιες ανάγκες πληροφορι... ανταλλαγής πληροφοριών. Σας ευχαριστώ πολύ, Διευθύντα. Ο κύριος Σερβίδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω λίγες ερωτήσεις, αυτές που έχουν να κάνουν με το πώς βλέπουμε το ρόλο του ΕΝΙΣΑ. Ε, ε, υπήρξε ένα ζήτημα, θύχτηκε το ζήτημα της θητείας, της σημερινής και πώς ε, εμφανίστηκε το σύστημα υπήρξαν πάρα πολλές ε, διαπραγματεύσεις και ιδίως με τη διεύρυνση περιπλάκησαν τα πράγματα γιατί υπήρχαν πολλά καινούρια νέα μέλη με διαφορετικές ε, προσδοκίες. Υπήρχαν κράτη που ήταν πολύ πίσω, άλλα που ήταν πολύ μπροστά. Ε, αυτά όλα δεν είναι καινούρια βέβαια, αλλά πιστεύω η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό ήταν ένα κοινωνικό πρόβλημα που υπήρχε εκεί στην έναρξη της σύστασης ε, του οργανισμού. Ε, θέλαμε να είμαστε πολύ σαφείς και να περιγράψουμε σαφώς τις αρμοδιότητες της ΕΝΗΣΑ για να περιορίσουμε κάθε παρέμβαση και να μπορούμε να είμαστε ο θεματοφύλακας αυτών των θεμάτων έναντι των κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα όμως θέλαμε να είμαστε και ανοιχτοί στις αλλαγές. Ο κόσμος αλλάζει και χρειάζεται διαρκώς καινούργια συνεργασία. Τα καλά νέα είναι ότι τα κράτη-μέλη το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Πιστε το Δεκέμβριο, ε, υιοθέτησε το Σεπτέμβριο ένα ψήφισμα σε συνέχεια του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένα ψήφισμα λοιπόν στη συνέχεια επίσης και της σχετικής συζήτησης ε, στην Ευρώπη για την ανάγκη συνεργασίας ε, στον τομέα της ε, ασφάλειας στην Ευρώπη. Χρειάζεται βέβαια περισσότερες χρειάζονται περισσότερες γνώσεις για την καλύτερη συνεργασία. Και υπό αυτήν την άποψη απίθυναν έκκληση και στον Ενίσα για να βοηθήσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σε σχέση με τις προτάσεις που, διατυπώνουμε, που διατυπώσαμε στις 30 Σεπτεμβρίου ε, δείχνει ότι θέλουμε και να συμπυκνώσουμε τις γνώσεις που ήδη υπάρχουν αλλά και να ε, συνενώσουμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, το χρήστη, τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη, όλους. Έτσι, θα Έτσι προσπαθούμε να διαμορφώσουμε και τον ρόλο για τον Ενίσα, να είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Και η, η, η, πρόκληση είναι να κάνουμε την Ευρώπη να αντιδρά ως μια ενιαία περιφέρεια. Και η Ευρώπη μπορεί να το κάνει αυτό γιατί έχει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και πρέπει να προσφέρει τη βοήθειά της. Χρειάζεται όμως τα αντίστοιχα εργαλεία. Ο Δόκτωρ Χέρμπρεχτ ήδη είπε ότι ότι έχουμε κάποιες πολύ βασικές ανάγκες ε, για τους χαράκτες πολιτικής, ε, τους οποίους πρέπει να βοηθήσουμε και για να τους βοηθήσουμε πρέπει να έχουμε τα καλά στοιχεία. Τι μπορώ πούμε, να σας πω για το 2010. Ε, έχω μια σειρά στατιστικών στοιχείων. Από πού προέρχονται, από πολιτές. Εντάξει, καλό. Μήπως όμως είναι διαπλεκόμενα τα συμφέροντά τους. Ασφαλώς και είναι διαπλεκόμενα. Όσο πιο ζωφερή η εικόνα, τόσο πιο πολλά λογισμικά και τεχνικά εργαλεία πουλούν. Ε, πρέπει αυτά να τα ξέρουμε. Κατά την προετοιμασία της δήλωσης πολιτικής μας έχουμε 80 σελίδες στατιστικά στοιχεία από τα οποία μπορεί κανείς ε, να αντλήσει, να συμπεράνει όποιο μήνυμα θέλει. Ε, νομίζω ότι για την ποινική πλευρά υπάρχει μεγαλύτερη κουλτούρα συνεργασίας φυσικά ε, βέβαια είναι δύσκολη η κατάσταση. Αν δούμε την άλλη πλευρά, δηλαδή τις παρολίγων επιτυχίες επιθέσεων, εκεί θα δούμε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, με τις αρμόδιες αρχές, τα στατιστικά γραφεία των κρατών μελών, για να έχουμε υγιή στατιστικά στοιχεία. Να μοιραζόμαστε όλοι επίσης τα στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να παρέχουμε αυτό που χρειάζονται οι χαράκτες πολιτικής, εσείς, οι κυβερνήσεις, αλλά επίσης στοιχεία που θα τα χρησιμοποιεί και ο ιδιωτικός τομέας. Σημαντικό είναι ο ιδιωτικός τομέας να λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση μια λογική ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου. Φυσικά χωρίς τους σωστούς πόρους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά με την μελέτη αντικτύπου βλέπει κανείς τις αναλύσεις που τεκμηριώνουν ε, ποιοι πρέπει να είναι οι οικονομικοί πόροι που χρειαζόμαστε. Οι χρηματοοικονομικές, οι δημοσιονομικές προοπτικές ακόμα δεν έχουν συζητηθεί και ολοκληρωθεί. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Και τέλος θα ήθελα να τα συνδέσω αυτά μεταξύ τους με μια πρόταση του ΕΝΙΖΑ για το συνολικό πλαίσιο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ατζέντα. Υπάρχει σημασία της ηλεκτρονικής ταυτότητας και της ηλεκτρονικής υπογραφής. Ε, πράγματι πρέπει να θεσπίσουμε και να εκπονήσουμε ένα πλαίσιο να βοηθήσουμε τη διαλειτουργικότητα αυτών των εργαλείων για να στηρίξουμε τις κυβερνήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και θα τελειώσω με τον πολίτη. Υπόθηκε ότι ο πολίτης πρέπει να είναι μέρος της εικόνας. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαμήρασης και Διάδοσης Στοιχείων πραγματικά έχει αποδέκτη και τον πολίτη και ο πολίτης είναι μέρος της πλατφόρμας ανταπόκρισης, απάντησης στο πρόβλημα. Αν δεν είναι ο πολίτης μέρος αυτού του συστήματος, δεν θα μπορούμε να τον έχουμε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Χάρτρικ θέλουν να απαντήσουν. Ο κύριος Γιάννης. Σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση, το συναγερμό ή την ανάγκη συγκέντρωση πληροφοριών θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε την έγκαιρη προειδοποίηση. Υπό το πρίσμα της αστυνομικής συνεργασίας έχουμε εφαρμόσει μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008 επί Γαλλικής Προεδρίας που πρόβλεπαν τη θέσπιση μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας προειδοποίησης. Αυτό υπάρχει σε δύο επίπεδα. Σε επίπεδο Europol, γιατί η Europol ε, λαμβάνει τις εκθέσεις των κρατών μελών, αλλά πρώτα για, να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να στείλουν τις εκθέσεις πρέπει να έχουν ήδη πλατφόρμες δικές τους. Έχουν όμως τέτοιες πλατφόρμες τα κράτη-μέλη. Έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες των κρατών μελών να καταγγέλουν ε, κυβερνοεγκλήματα, εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, γιατί δεν διαθέτουν όλα τα κρατημέλη τέτοιες πλατφόρμες και εμείς ε, στηρίζουμε και οικονομικά τις χώρες προκειμένου να ε, εγκαινιάσουν τέτοιες πλατφόρμες. Υπάρχουν ήδη hotlines, ανοιχτέ γραμμές και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε κάποιες ε, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις Μπορούν όμως οι πολίτες πολύ γρήγορα να καταγγέλουν spam phishing ή ε, παράνομο περιεχόμενο. Δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες τέτοιες δυνατότητες. Η Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα Προειδοποίησης ε, ήδη ασκεί από αυτήν την άποψη μια πίστη στα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν τέτοιες δομές να τις επισπεύσουν. Είχαμε και τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Απριλίου επί Ισπανική Προεδρίας. Εκεί υπευλήθη μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν να αξιολογήσει κατά πόσο θα μπορούσε να, να ιδρύσει ένα κέντρο εγκλήματος του κυβερνοχώρου. Δηλαδή να συγκεντρώσει τι τις διάφορες πληροφορίες από κράτη-μέλη, από ιδρύματα κτλ. ώστε να διευκολύνει τις έρευνες και τη συλλογή πληροφοριών για θέματα απειλών του κυβερνοχώρου. Η ανταλλαγή των πληροφοριών κατά τη γνώμη μας έχει κέρια σημασία, έχει νευραλγικό ρόλο και σημειώνουμε αρκετή πρόοδο εκεί. Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους, φυσικά η οδηγία δεν καλύπτει το στρατιωτικό τομέα, αφορά το πολιτικό σκέλος και απευθύνεται κυρίως στα κράτη-μέλη, αλλά ο διαχωρισμός μεταξύ του στρατιωτικού και του μη στρατιωτικού τομέα είναι όλο και πιο ασαφής και στενή η διαφορά. Στα πλαίσια της ε, υποβολής εκθέσεων έχουμε λάβει καταγγελίες κάποιων ε, στρατικών αεροσκαφών που έμειναν καθυλωμένα στο έδαφος επειδή τα συστήματά τους ε, προσβλήθηκαν από botnet, από τέτοιο ιό ή από ιό μέσω κλειδιού μνήμης, USB. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα με τον Ανδρέα Σερβίδα συμμετείχαμε σε μία άσκηση που έγινε στις Πολιτείες κατά κυβερνοαπειλής και στι Ηνωμένε Πολιτείε εκεί συμμετέχει και ο στρατός, γιατί και ο στρατός λαμβάνει πληροφορίες για το πώ έλαβε χώρα η, η απειλή αυτή, πώς πραγματοποιήθηκε μάλλον η απειλή και ούτω καθεξής. Και στο μέλλον όλοι φυσικά οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν σε τέτοιε ασκήσει. οπότε ο συντονισμός είναι απαραίτητο και με το στρατό, κάτι που δεν ισχύει μέχρι στιγμή. Δεν αποκλείεται όμω να συμβεί στο μέλλον και μάλλον αργά ή γρήγορα θα είναι κάτι αναπόφευκτο. Αλλά είναι και ευαίσθητο θέμα εξαιτία ε, του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών των πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του ΕΝΙΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλεια Δικτύου και Πληροφοριών, είναι φυσικά σημαντικό και είναι σημαντικό και ο ρόλο τη Europol. Σα μίλησα για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Προειδοποίηση. σω η Europol θα ήταν ο καλύτερο υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πάταξη του Κυβέρνου Εγκλήματος και αν θέλουμε μια συνολική αντίδραση απέναντι στο έγκλημα θα πρέπει να, εφοδιάσουμε, να εφοδιαστούμε με τα απαραίτητα μέσα. Και σίγουρα μια πρόταση που θα κατατεθεί θα πρέπει να την εξοπλίσουμε με τα κατάλληλα μέσα, με καλύτερο συντονισμό μεταξύ των, της Europol, της Eurojust, του CEPOL, της του ENISA, γιατί και η ΣΥΠΟΛ συμμετείχε στην κατάρτιση των διοκτικών αρχών, για παράδειγμα. Και η Europol, παρόλο που δεν έχει ω πρωταρχική τη αποστολή αυτό το έργο τη κατάρτιση τέτοιες δραστηριότητες. Οπότε έχουμε πολλού οργανισμού, πολλέ υπηρεσίε και διαφορετικού ρόλου, Ίσως θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το συντονισμό μεταξύ του. Σε ό,τι αφορά την υφαρπαγή ταυτότητα και την απάτη με τέτοιου είδου υφαρπαγή ταυτότητα, έχουμε να θέσει μία μελέτη σε μία εταιρεία προκειμένου να εξετάσει αυτό το θέμα της υφαρπαγής ταυτότητας και της συναφούς απάτης. Μάλιστα έγινε ήδη μια δεύτερη ακρόαση με αυτό το θέμα με κοινή οργάνωση Επιτροπής και Βελικής Προεδρίας. Και θα ακούσουμε σύντομα τα απορίσματα αυτής της, την έκβαση αυτής της ακρόασης. Τέλος, συμφωνώ ως προς την ευθύνη. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ευθύνη των χρηστών για προστασία των υπολογιστών τους. Γιατί στα αυτοκίνητα έχουμε τις ζώνες ασφαλείας και ξέρουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις συνδέσουμε. Αλλά και οι παραγωγοί λογισμικού έχουν υποχρέωση το λογισμικό τους να είναι όσο πιο ασφαλές γίνεται. Τώρα που θα βρούμε την ισορροπία μεταξύ των χρηστών και των παραγωγών. Είναι αρκετά λεπτό το θέμα, αλλά ίσως ε, έχουμε μιλήσει αυτό το θέμα της προσωπικής ευθύνης των χρηστών. Αν ζητήσω όμως από τους χρήστες να αναλάβουν την προσωπική ευθύνη, θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να μας κοινοποιήσουν τα προβλήματα. Και άρα όλες οι χώρες θα πρέπει να εφοδιαστούν με τέτοιες πλατφόρμες που να δίνουν δυνατότητα στους πολίτες να καταγγέλουν τέτοια φαινόμενα. Εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κάτι πολύ μικρό για το θέμα της στατιστικής που Κοιτάξτε, πρέπει να έχετε κατά νου. Ας πάρουμε ας πούμε την περίπτωση μιας ε, κυβερνοεπίθεσης. Κατ' ουσίαν έχουμε και πάλι δύο θέματα. Έχουμε το θέμα της ασφάλειας, ε, του δημόσιου φορέα που δέχεται την επίθεση και Προφανώς θέλει το σύστημα των δυνατών τα συστήματα του να λειτουργήσουν. Πρέπει λοιπόν να αξιολογηθεί η ζημιά και να λειτουργήσει και πάλι το σύστημα. Και μετά υπάρχει και το ποινικό στοιχείο. Ε, προφανώς ε, θα υπάρχει ενδιαφέρον να διωχθεί αυτό το έγκλημα και γι' αυτό εσείς πρέπει να κρίνετε κατά πόσον όλες αυτές οι υποθέσεις θα φτάνουν τελικά σε ιδιοκτικέ αρχές γιατί ενδέχεται ορισμένες υποθέσεις για χι να μην αναφερθούν καν στις διοκτικές αρχές. Όσον αφορά τώρα ε, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος, επειδή υπενικτήκατε λιγάκι το θέμα της ε, εκπαίδευσης, προφανώς η εκπαίδευση είναι ένα καθοριστικό στοιχείο έτσι ώστε τα δικονομικά να ε, είναι αντικείμενο εκπαίδευσης και γενικότερα η εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες. Νομίζω ότι κατονούμε τώρα όλοι περί τίνος ε, πρόκειται. Δεν ε, είναι τα σπάμ και τα κακόβλα email που έχουμε καθημερινά. Θυμάμαι μια περίπτωση από την Πολωνία όπου έγινε επίθεση στο επίσημο website του πρόεδρου της Πολωνίας και αυτό ήταν μάλιστα πολύ αστείο γιατί όσοι έμπεραν σε αυτό το website ε, διοχετεύονταν σε κάποιο άλλο ε, το οποίο μερικοί δημοσιογράφοι επειδή είχε σχέση με πορνογραφικό υλικό ορισμένοι δημοσιογράφοι ε, το χαρακτήρισαν πιο ενδιαφέρον. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή δεν είναι η τελευταία μας ε, συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Λυπάμαι πάρα πολύ που το Συμβούλιο αρνήθηκε να συμμετάσχει, αλλά θα έχουμε ε, σε δύο μέρες την ευκαιρία να κάνουμε ερωτήσεις ε, στην Βαρόνη Άστον, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση για την κυβερνοασφάλεια. Εγώ λοιπόν προτείνω να συζητηθεί το θέμα στους ε, συντονιστές Ίσως ε, μπορούμε να προτείνουμε στην ε, ΑΦΕΤ να υποβάλει μια προφορική ερώτηση στην Κομισιόν και το Συμβούλιο σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις χώρες μας και πώς πρέπει να αντιδράσουμε στο ενδεχόμενο της επίθεσης. Είναι σοβαρό το θέμα γιατί γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ γίνεται αυτή η συζήτηση ε, κατά πόσον αυτή η κυβερνοεπίθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του άρθρου 5 ή όχι. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να το συζητήσουμε στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ και όλους